Κυρίες και κύριοι, ε, σας παρακαλώ να λάβετε θέση για να μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Πάμε λοιπόν στην έκθεση ζήμων για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ε, ποιο είναι παρακαλώ υπέρ. Dagegen. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε, προχωράμε. Τροπολογία 149, τροποποιημένη, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κυρία Βόρτμαν Κόλ παρακαλώ. με βάση το άρθρο 2, τροπολογία 154, ε, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 42 της Επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές, 151 θεωρημένη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 72 μέχρι 74 της Επιτροπής ε, καταπίπτουν 155 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται Συγγνώμη λέει ο πρόεδρος απορρίπτεται Σας ζητώ συγγνώμη 151 αναθεωρημένη υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται όμως τώρα. 152 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε τώρα ε, στην τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής με ονομαστική ψηφορία, η οποία και αρχίζει παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα παρακαλώ. Α, da Εγκρίνεται. Λοιπόν, ε, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε, έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Ζήμων. Πάμε τώρα στην έκθεση του συναδέλφου Βον, ε, κατευθυντήριε γραμμέ για τον προπολογισμό. Η τροπολογία υπαριθμών 7 αποσύρθηκε στη 2 ονομαστική ψηφορία. Άρχεται η ψηφορία. Έκλεισε. Εντάξει, ας μείνει λίγο ακόμα ανοιχτή. Ψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Έκλεισε τώρα η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Προχωράμε στην παράγραφο 9. Υπέρ παρακαλώ. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 με ονομαστική ψηφοφορία. Ε, ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 8 η οποία αποσύρθηκε. Η τροπολογία υπαριθμών 3 υπέρ παρακαλώ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι πέντε με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία υπερθμών 6. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα και ψηφίζουμε για το σύνολο του ε, κειμένου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Βόν. Επόμενο θέμα, πολιτές πρόγραμμα για το δυτικό απόθεμα Σαφριδιού. Ε, ποιος συμφωνεί παρακαλώ με την τροπολογία υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα ε, στην συμβολή της κοινή αληθικής πολιτικής στην παραγωγή δημοσίων αγαθών. Έχουμε πρώτες ψηφίσματος από πολλές πολιτικές ομάδες. Ε, ε, καταρχήν, ε, παράγραφος 23 του αρχικού κειμένου. Ε, ψηφίζουμε σε τμήματα. Υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έλεγχο θέλετε. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το σύνολο του κειμένου. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στο ψήφισμα για τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία. Ο κύριος Μπάτεν ζήτησε το λόγο. Κύριος Μπάτεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι η πρώτη τροπολογία στην έκθεση αυτή νομίζω ότι δεν ήταν ε, στην ιστοσελίδα σήμερα το πρωί, αλλά έπρεπε να υπάρχει για να μπορούν να τη δουν οι συνεργάτες μας, οι οποίοι προετοιμάζουν τον κατάλογο ψηφοφοριών πρώτη φορά φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο από ό,τι μου λένε. Τουλάχιστον αυτή είναι η εμπειρία, η πενταετής εμπειρία των συνεργατών που προετοιμάζουν τις λίστες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν ε, οι συνάδελφοι. Θέλω να το προσέξετε ότι αν ψηφιστεί αυτό καταπίπτει όλη η υπόλοιπη έκθεση θα μπορούν οι Ούγγροι να, ορίζουν τα του συντάγματό χωρίς χωρί καμία πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να διαξαγάγεται έρευνα. Γιατί δεν φαίνεται σωστά ο κατάλληλο ψηφοφοριών. Κύριε Μπάτεν, για ποια τροπολογία ένα μιλάτε, για ποια πρόταση ψηφίσματος. Για την πρώτη είναι η τροπολογία του ΕΛΚΑ, ε, για αυτήν ψηφίζουμε. Εσείς μίλησατε για ψήφισμα του ΕΛΚ. Εντάξει, το καταλάβαμε, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα, ε, θα ε, ψηφίζουμε για τις προτάσεις ψηφίσματος ως έχουν κατατεθεί. Και γι' αυτό ψηφίζω, ψηφίζουμε πρώτα για το πρόταση ψηφίσματος του ΕΛΚ. Πρόταση ψηφίσματος του ΕΛΚ. Ε, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μισό λεπτό. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Από ό,τι φαίνεται ναι ε, και έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα ε, ψηφίζουμε για την τροπολογία του, για το ψήφισμα του ΙΣΕΑΡ ε, της ομάδας ε, των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών υπέρ κατά αποχές η ίδια ψηφοφορία, η ίδια πλειοψηφία, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ε, ψήφισαν όλοι. Ωραία, έκλεισε η ψηφοφορία. Η ίδια η πλειοψηφία απορρίπτεται. Τώρα, στην πρόταση ψηφίσματος τεσσάρων πολιτικών ομάδων, Καταρχήν ψηφίζουμε για την τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται. Τώρα ε, ψηφίζουμε για το αρχικό κείμενο της παραγράφου 3. Με ονομαστική ψηφοφορία. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην παράγραφο 4 που θα ψηφίσουμε σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παράγραφος 4 πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε λοιπόν η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για την τροπολογία υπαρτιμών 4 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πολύ ωραία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στο αρχικό κείμενο της παραγράφου υπαριθμών 7. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Υπέρ. Όχι, λάθος λέει ο πρόεδρος. Ε, ψηφίζουμε τώρα. Άρχεται η ψηφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πολύ ωραία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για το σύνολο αυτού της πρώτης ψηφίσματος υπέρ κατά αποχές ε, για να είμαστε σίγουροι ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Η πρόταση εγκρίνεται. Kommen nun Πάμε τώρα στην κατάσταση στη Ρωσία. Πρόκειται για κοινή πρόταση ψηφίσματος από πέντε πολιτικές ομάδες. Ψηφίζουμε για την πρώτη παράγραφο υπέρ κατά αποχές. Δεν βλέπω. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε για την παράγραφο 15 του αρχικού κειμένου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για το σύνολο του σχεδίου ψηφίσματος. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Νομίζω ότι τώρα Πάμε στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Μαρόκου σχετικά με δύο μετρά ελευθέρωση για γεωργικά προϊόντα και προϊόντα. Πάμε στο... στην κοινή πρόταση ψηφίσματος ε, των Πρασίνων και της ε, Γκουε με ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται η πρόταση. Πάμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος των πρασίνων παρακαλώ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτή η πρόταση. Πάμε τώρα στην κοινή πρόταση ψηφίσματος τεσσάρων πολιτικών ομάδων. Ψηφίζουμε για την τροπολογία υπαρτιμών 4 σε ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5, επίσης με ε, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 1 αλλά μου έχουν πει ότι η κυρία Μουσκαρντίνη επιθυμεί να καταθέσει προφορική τροπολογία. Σωστό, κυρία Μουσκαρδίνη. Ναι, πρόεδρε ρωτώ κατά πόσον είναι δυνατόν στην τροπολογία υπαρτμών 6 στο τέλος της παραγράφου μετά από εκεί που λέει Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσθέσουμε εάν η αξιολόγηση αντικτύπων αποδείξει αντικειμενικές δυσκολίες στους τομέους που συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία τότε η Επιτροπή πρέπει αυτό να το λάβει υπόψη της αναθεωρώντας την κοινή γεωργική πολιτική και αυτή την ε, τροπολογία την καταθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες του γεωργικού τομέα. Πρόεδρος, ε, πρέπει να ερωτήσω ε, κατά αυτής της ε, προφορικής τροπολογίας αν σηκωθούν 40 συνάδελφοι και σηκώθηκαν πάνω από 40. Λυπάμαι κύριε Μουσκαρδίνη, απορρίπτεται η προφορική σας τροπολογία και τώρα ψηφίζουμε για την τροπολογία 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 1. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 2. Ψηφίζουμε ονομαστικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έτσι λοιπόν, καταπίπτει το αρχικό κείμενο και πάμε τώρα στην τροπολογία 6 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα πάμε στην τροπολογία Τρία με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε ε, για το σύνολο του κειμένου υπέρ παρακαλώ. Ποιος συμφωνεί με το κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για την έκθεση του συναδέλφου Μπουβί με ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ κύριε Μπουβί. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα μακρηγορήσω. Θέλω να πω απλά ότι η έκθεση για την ε, συμφωνία ε, που φέρει το δικό μου όνομα και επειδή υπήρχε συμφωνία στο πλαίσιο τη Επιτροπή δεν Εμπορίου που ήταν υπέρ τη συμφωνία, ναι, εξακολουθεί να φέρει το όνομά μου η έκθεση, αλλά σα ζητώ να ψηφίσετε κατά τη έκθεση. Να βάλετε όχι. Όσοι είστε κατά τη συμφωνία, να ψηφίσετε όχι στην έκθεση. Να καταψηφίσετε την έκθεση. Ευχαριστούμε κύριε Μπουβή για αυτή τη διευκρίνηση. Ψηφίζουμε τώρα για την έκθεση του συναδέλφου Μπουβέ. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφορία. Εγκρίνεται η έκθεση. Παρακαλώ κύριε Μπόβε. Μετά και το αποτέλεσμα υποκλίνομαι ε, στη σοφία της πλειοψηφίας ε, και αποσύρω το όνομά μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν ε, σε αυτή τη συζήτηση γιατί πιστεύω ότι για πρώτη φορά έγινε μια συζήτηση για το διεθνές εμπόριο και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συζητήσεις που έγιναν. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μποβέ απέσυρε το όνομα του, ε, άρα υποθέτω με την πρακτική που ακολουθούμε θα μετατραπεί αυτό σε έκθεση Μορέρα. Ε, συγχαρητήρια κύριε Μορέρα. Πάμε τώρα στην κατάσταση στη Συρία. Κοινή πρόταση ψηφίσματος από πέντε πολιτικές ομάδες. Ψηφίζουμε για το σύνολο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19η Σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Ε, ψηφίζουμε για την 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 4 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι 7 υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πολύ ωραία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 9 και 21 είναι οι ταυτόσημες, ε, γι' αυτό λοιπόν ψηφίζουμε και για τις δύο ονομαστικά ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 με ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξανά από την αρχή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 16 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το αρχικό ε, κείμενο προφορική τροπολογία του κυρίου Πρέντα. Κύριε Πρέντα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ja, bitte, Sie haben das Wort. Έχετε λόγο κύριε Πρέντα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας uh, προτείνω το πρώτο τμήμα της uh, παραγράφου 29 να διαγραφεί εκεί που λέει καταδικάζει και τα υπόλοιπα μέχρι τη χρήση της uh, θανατικής ποινής και αυτό για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Το απόγευμα θα ψηφίσουμε για ένα ψήφισμα το οποίο αφορά ακριβώς αυτό το θέμα. Και αυτή η πρόταση ψηφίσματος ε, που θα ψηφίσουμε το απόγευμα είναι πολύ καλύτερη από αυτή που ψηφίζουμε τώρα. Υπέρ, λέει ο Πρόεδρος. Υπέρ αυτό που προτείνει ο κ. Πρέντα. Κατά, κατά. είναι κανείς κατά αυτής της προφορικής τροπολογίας. Ε, εντάξει, τέλειωσε τώρα. κατέπεσε η προφορική τροπολογία, ε, παραμένει έχει 29 γιατί 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 31 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζουμε. Για την 33 ε, αρχικό κείμενο ε, δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε έκλειση ψηφορία. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Για το αρχικό κείμενο της παραγράφου 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του κειμένου υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενο θέμα. Η πρόσβαση των τυφλών στα βιβλία. Είναι ε, πρόταση της Επιτροπής Αναφορών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περιφερειακή Σύμβαση για Πανευρομεσογειακούς Προτιμησιακούς Κανόνες Καταγωγής. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για το σύνολο του κειμένου υπέρ. Κατά. Η ονομαστική ψηφορία είναι για την επόμενη έκθεση. Εδώ δεν προβλέπεται ονομαστική ε, έκθεση. Γι' αυτό λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην έκθεση Μενέντες Valle, ε, το ίδιο θέμα, ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφορία. Εγκρίνεται, συγχαρητήρια. Και τώρα έχουμε μόνο να ψηφίσουμε για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παρακολούθησης της Γης. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πολύ.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 Panie i Panowie Posłowie, rozpoczynamy procedurę. Παρακαλώ, μπορούμε